Όπως γνωρίζετε κυρίες και κύριοι, η διάσκεψη των Προέδρων των πολιτικών ομάδων αποφάσισε ε, να ακυρωθεί η μήνυ σύνοδος ε, των Βρυξελών τον Νοέμβριο. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ε, εν συντομία επευκαιρία. Όπως γνωρίζετε, στις Βρυξέλλες απέκτησε αστάθεια η οροφή του ημικυκλίου. Κάνουμε ε, συχνά επιθεωρήσεις ε, και είδαμε ότι από τις 23 δοκούς οι τρεις έχουν ρογμές και με ενημέρωσαν τον Αύγουστο ότι αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο και γι' αυτό ε, αποφάσισα αμέσως να κλείσει η αίθουσα της Ολομέλειας στις Βρυξέλλες. Η πρώτη γνωμάτευση που μας υπευλήθη προέβλεπε μάλλον είχε ε, διαπιστώσει ότι η πιο επικίνδυνη θέση ήταν θέση του Προέδρου στην Ευρωπα... στο ημικύκλιο. Οπότε καταλάβατε ότι το έκλεισα αμέσω στο ημικύκλιο. Ε, οι επόμενες ε, επιθεωρήσεις έδειξαν ότι πρόκειται για σοβαρή ζημία που δεν έχει να κάνει με πλημελή κατασκευή, με κακοτεχνίες ή αδυναμία υλικού από ό,τι φαίνεται πρόκειται για φθορά του υλικού που δεν ε, μπορούσε να είχε προβλεφθεί. Παρακάλεσα το Γενικό Γραμματέα ε, να συμβουλευθεί όλους τους εμπειρογνώμονες και τη βελγική κυβέρνηση. Ε, ενημέρωσα και τον Πρωθυπουργό κύριο Ντερούπο. μας έχει διαθέσει εμπειρογνώμονες από την αντίστοιχη υπηρεσία κτηρίων, για να μας βοηθήσουν θεωρούμε ότι θα χρειαστεί κάποια περίοδος αρκετά μακρά για την επισκευή. Πρέπει να σας πω ότι χρειάστηκε να ρίξουμε την, την ε, οροφή, μάλλον, συγγνώμη, ναι. για να μην πέσει να τη στηρίξουμε με, με ε, σκαλοσιές. Αλλά είναι τόσο βαριές αυτές οι σκαλοσιές που πιέζουν και το δάπεδο ε, και χρειάστηκε να εκενώσουμε και τα γραφεία και τους χώρους που βρίσκονται κάτω από την Ολομέλεια ε, που έχουν καταστεί πλέον άχρηστοι προς το παρόν γι' αυτό έχει αποκλειστεί όλη αυτή η πτέρυγα. Ε, το επόμενο διάστημα θα συμβουλευτούμε και δύο Ινστιτούτα Διεθνούς Κύρους και Φήμης. Τώρα το πότε θα ξανανοίξει το ημικύκλιο στις δεν γνωρίζω. Αλλά σύμφωνα με την εμπειρία χρειάζονται το χρόνο τους τέτοιες εργασίες έτσι, οικοδομικές. Παρά τις δύσκολες αυτές συνθήκες συνεχίζονται οι εργασίες μας και παρόλα αυτά ενημέρωσα και την ε, καγκελάριο κυρία Μέρκελ και την κάλεσα στο Κοινοβούλιο σε ανοιχτή δημόσια διάσκεψη των Προέδρων γιατί θα ερχόταν το Νοέμβριο η κυρία Μέρκελ στην Ορομέλεια και οποία έκπληξη στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μας παραχωρεί την αίθουσά του που είναι και μεγαλύτερη μετά την Ολομέλεια για να υποδεχθούμε και την κυρία Μέρκελ. Εκεί θα συνεδριάσει δημόσια η διάσκεψη των Προέδρων και ουσιαστικά η διαδικασία θα είναι σαν είναι η Ορομέλεια. Το ε, συνεννοήθηκα και το συμφώνησα αυτό και με την κυρία Μέρκελ την ίδια. Θυμίζω κάτι σύντομα. Δεν ξέρω τους τελευταίους μήνες πόσες φορές σας έστειλα επιστολές που ελπίζω να τις διαβάσατε όλες. για μια φωτογραφία που θα βγάλουμε αύριο στις 12.30 λίγο πριν τις ψηφοφορίες θα έχουμε μια πανοραμική ε, φωτογραφία σε ποιότητα τρισδιάστατη, 360 μοίρες με τους βουλευτές στα έδρανά τους. Θα θυμάστε γιατί σας το έχω ε, ε, στείλει επανειλημμένα σε επιστολή, σας έχω περιγράψει. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που ισχυρίζονται ότι δεν πήραν ποτέ τέτοιο γράμμα. Δεν το πιστεύω. Μάλλον δεν το διάβασαν. Πάντως, για όσους δεν έχουν δει τις σειρίδες τους, για λόγους πρακτικούς ή άλλου, ε, θυμίζω ότι αύριο, λοιπόν, 12 και 25, εδώ θα κάνουμε μια φωτογραφία λήψη 360 μοίρων και θα το βάλουμε στο διαδίκτυο για να μπορεί κάθε ψηφοφόρος και κάθε ενδιαφερόμενος να εντοπίζει αμέσως τον κάθε βουλευτή. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ερχόμαστε τώρα στη συζήτηση για το Γενικό Προεπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013. Όλα τα τμήματα. Θα δώσω λοιπόν το λόγο πρώτα στον κύριο Τζοβάνι Λαβία, τον εισηγητή μας. Έχετε το λόγο. Presidente, Ministro Mauro Κύριε Μαυρογιάννη, Πρόεδρε και Επίτροπε Λεβαντόφσκι, με την αυριανή ψηφοφορία